Καλησπέρα. Να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη. Και μετά να κάνω και τις ανακοινώσεις. Να ξεκινήσουμε το εποπτικό μας έργο. Και θα έρθει και ο εισηγητής. Πρώτον, είχαμε στις 24 Μαΐου συνάντηση ΕΚΟΝ-ΑΦΚΟ μάλλον θα γίνει στις 24 το πρωί για να εξετάσουμε τις τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της ε, ΕΚΤΑΦ. Έχουμε ε, επίσης τη συνόψη των αποφάσεων των ε, συντονιστών. Έχουμε τον ορισμό εισηγητών γνωμοδοτήσεων και για τα άλλα θέματα αναφέρονται εκεί στη συνόψηση των αποτελεσμάτων Τη συνεδρίαση των συντονιστών. Α, όχι, οι τελευταίοι δεν έχουν γίνει. Οικονομική διακυβέρνηση. Θα συναντηθούμε με το Eurogroup, τους υπουργού Οικονομικών μια σειρά κρατών μελών, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Αυστρία, σε μια συνάντηση στις 12 Ιουλίου για το πακέτο για την Οικονομική Νομισματική Ένωση και θα ζητήσουμε και ενδιάμεση έκθεση για το, με βάση το κανόνα 99.5 για το ESM και το EMF και θα έχουμε το αντελικό κατάλογο των ε, ορισμών και είδατε και το σχέδιο της προφορικής ερώτησης προς την Κομισιόν έχει διανεμηθεί για μια ζήτηση στην Ολομέλεια για την ΟΝΕ και συνέχιση του καθεστώτος του Eurostat. Θα στείλουμε μια επιστολή στο Γενικό Διευθυντή της Eurostat ζητώντας μία γραπτή δήλωση για την εφαρμογή του στατιστικού προγράμματος. Επίσης αποφασίστηκε ότι θα καλέσουμε τον πρόεδρο του, ε, της ομάδας εργασίας για το Eurogroup όπως κάναμε και στο παρελθόν το σχέδιο προγράμματος για την αποστολή στην Αθήνα στις 25-26 Ιουνίου θα σταλεί στους συντονιστές και θα υπάρχουν τέσσερις ε, από το ΕΛΚ, τέσσερις από τους σοσιαλιστές και ένας από τους άλλους. Ο κύριος Στολογιάν θα είναι ο εισηγητής και οι ε, σκιώδεις θα είναι επίσης ε, αρμόδιοι. Ο τίτλος και το χρονοδιάγραμμα συμφωνήθηκε. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στις 30 Μαΐου, θα ψηφιστεί 18-19 Ιουνίου στην ΕΚΟΝ, τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Θα καλέσουμε τον πρόεδρο του ΕΦΡΑΓ για ανταλλαγή με τα μέλη της ΕΚΟΝ, αντιπροσωπείες και επισκέψεις. Είπαμε ότι η θέση για την ΕΚΤ της ΓΚΟΕ δεν θα πάει σε άλλον. Δεύτερο εξάμεινο αποστολές θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα DONT για τις αποστολές της ΗΠΑ τον Ιούλιο εφόσον πάρει απόφαση η διάσκεψη των Προέδρων για το πόσοι θα πάνε. Αν είναι 7, 3 ΕΛΚ, 3 σοσιαλιστές, 1 CCR. Αν είναι 8, θα προσθεθεί και ένας ΑΛΔΕ. Αν είναι 9, 4 ε, ε, ΕΛΚ, 3 σοσιαλιστές, 1 CCR, 1 ΑΛΚΕ. Προπαρασκευή για το τέλος της θητείας αποφασίσαμε ότι ανάλογα με το χρόνο που θα έχουμε θα κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων στο τέλος της Προεδρίας για 30-40 λεπτά ή καθόλου. Και η εποπτεία θα γίνει μόνο αν υπάρχει επίγουσα ανάγκη για κάποιο θέμα. Δεν θα έχουμε έκτακτες συνεδριάσεις κατά τις ε, τυρκουάς 38, 44 και 51 δηλαδή, και τις Δευτέρες στο Στρασβούργο και την Πέμπτη το απόγευμα κατά την εβδομάδα των ομάδων θα, χρησιμοποιήσουμε, θα χρησιμοποιούνται μόνο εάν δεν γίνεται να αποφευχθεί. Επίσης θα καλέσουμε τον πρόεδρο της υψηλού επίπεδου Task Force για τις επενδύσεις στην κοινωνική υποδομή σε μια ανοιχτή συνεδρίαση των συντονιστών για την παρουσίαση της έκθεσης για να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις για τις κοινωνικές υποδομές και συμφωνήσαμε μετά από αίτημα του συντονιστή του ECR να υπάρξει μια περίοδος εποπτείας. Α, όχι, όχι, όχι, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, είναι θέμα της ημερήσης διάταξης. Δεν έχει αποφασιστεί. Σημείο 3. Ε, τι έγινε στους τριμερείς διαλόγους. Ο δεύτερος ε, τέτοιος διάλογος για το κανονισμό BAS έγινε στις 14 Μαΐου. Α, όχι, δεν είναι κανονισμός, είναι οδηγία. Πολύ επικοδομητικός. Οι διαπραγματευτές κατέληξαν στο άρθρο 3 εγγυήσεις 4 ανεξαρτησία του NCA και 5 πόροι 12 υπολογισμός των προστήμων 22 ε, ασυλία για φυσικά άτομα και συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το υπόλοιπο κείμενο. Η ομάδα μας παρουσίασε τη θέση της για το άρθρο 21 συνοπτικές ε, αιτήσει και το πακέτο επίοικιας για την επόμενη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου στις 30 Μαΐου. Τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την περίοδο εποπτείας για τη φερικαιότητα 2, όπως ξέρετε. Πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπω τον κύριο Κλίντς. Χαίρομαι που είστε εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείτε να εκπροσωπήσετε τον εισηγητή του ΕΛΚ. Οπότε να σας διασκεδάζω, να σας διασκεδάσω εξηγώντας ε, γιατί εισήχθη αυτή η περίοδος εποπτείας και ελέγχου για να βελτιώσουμε τον έλεγχό μας για τα μέτρα επίπεδου 2 που είναι τόσο σημαντικά και αποφασίσαμε να συζητήσουμε και να ελέγξουμε το θέμα φερεγγιότητα 2 δεν σας εκπλήσει και είναι εξελίξει η εξέταση του τόσο σημαντικού αυτού θέματος αυτής της κατεξοδότησης πράξης για τις απαιτήσει, ε, κεφαλαιακές απαιτήσει φερεγγιότητας και η ευρύτερη επανεξέταση και χαίρομαι που έχουμε τον Φάουστ Παρέντε, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΙΟΠΑ και τον κύριο Μερλά που είναι ο Διευθυντής Τη γενική Διεύθυνση ΦΙΣΜΑ για τις ε, χρηματαγορές. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε. Λοιπόν, ΕΙΟΠΑ. Ο κύριος Φάουστο Παρέντε. Η ΕΙΟΠΑ μας έδωσε τεχνικές συμβουλές για το θέμα αυτό. Έχουμε εδώ τον κύριο Παρέντε. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Μερλέ. Σας ε, καλωσορίζω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βεβαίως να συμβάλλουμε σε αυτή την ε, λειτουργία ελέγχου. Η Φεργιώτα 2 λειτουργεί τώρα δύο χρόνια. Και τώρα θα πρέπει να γίνει μία ε, κάποια συντήρηση για να βελτιώσουμε το σύστημα. Δίνουμε τεχνικές συμβουλές για την Κομισιόν, πρόσφατα τα δώσαμε, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά τους, ασχοληθήκαμε με τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι η περισσότερη χρήση της αρχής της αναλογικότητας. Δεύτερον, ε, να καταργηθούν οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Να βοηθήσουμε δηλαδή την ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Και το τρίτο είναι να καταργηθούν ορισμένε τεχνικές ασυνέπειες. Όπως θα είδατε, οι συμβουλές μας είναι μακροσκελής. Εγώ θα ασχοληθώ με μερικά κύρια σημεία. Τώρα για την αναλογικότητα. Έχουμε προτείνει, έχουμε προτείνει προς την Κομισιόν να κάνει κάποιες απλουστεύσεις για κάποιους υπολογισμούς, για, κάποιους, ε, για κάποια υποστοιχεία των κινδύνων Βεβαίω όλα αυτά είναι προαιρετικά. Για να καταλάβουν ε, οι επιχειρήσεις του κλάδου εάν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν. Επίσης, δεν πρέπει να εξαρτώμεθα τόσο πολύ από εξωτερικούς οργανισμούς ε, πιστοληπτικής ικανότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας και και θα πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμόσουμε την προσέγγιση διαφάνειας όταν κάποιοι επενδυτές επενδύουν σε συλλογικούς ε, επενδυτικούς φορείς. Δεύτερον, πώς θα συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και εδώ θέλουμε κάποιες απλουστεύσεις στην αντιμετώπιση ε, του μη αξιολογηθέντος χρέους και, της μη, και των μη ε, εισηχθέντων τίτλων. Αυτό το κάναμε και στο παρελθόν για τις επενδύσεις υποδομών. Εντοπίσαμε κάποια αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλιστές να αξιολογήσουν τον κίνδυνο αυτών των επενδύσεων. Παρόμοια με αυτό που κάνουν για ε, τους αξιολογηθέντες και εισηγμένους τίτλους. Είναι αντικειμενικά αυτά τα κριτήρια, αλλά σε ένα βαθμό εξαρτώνται από την κρίση και την πείρα των ε, ασφαλιστών. Ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λοιπόν. Και επειδή έχει περάσει κάποιος χρόνος, έχουμε αναθεωρήσει και κάποιες σταθμίσεις. Για παράδειγμα, τους κινδύνους θεομηνιών, ε, βοήθεια και ιατρικές δαπάνες. Ε, κάποιες ειδικέ ε, πλευρές ε, των ασφαλίσεων που από καιρού εις καιρών πρέπει να επαναξιολογούνται από πλευρά στάθμισης ή βαθμονόμησης. Επίσης του λέμε να ανασταθμίσει τον κίνδυνο από τα επιτόκια. Γιατί αυτά που είδαμε πρόσφατα δεν μπορούσε να προβλεφθεί όταν καθορίστηκε παλιότερα η προσέγγιση μας. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες επαναβαθμονομήσεις. Είναι τμήμα των συμβουλών που συζητήσαμε με τις επιχειρήσεις και τους άλλους ε, ενδιαφερόμενους. Οι επιπτώσεις τώρα των προτάσεών μας μπορεί να είναι σημαντικές. Γι' αυτό προτείνουμε η νέα μεθοδολογία να εισαχθεί σταδιακά ε, κατά τη διάρκεια μιας περίοδου τριών ετών. Κάτι επίσης σημαντικό. Η αντιμετώπιση και ο τρόπος χρήσης που αξιοποιείται η δυνατότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλόμενων φόρων. Μετά από δύο χρόνια είδαμε πώς αξιοποιείται αυτό το στοιχείο και διαπιστώσαμε ότι 70% του ποσού αυτού του στοιχείου των ισολογισμών εφαρμόζεται με παρόμοιο τρόπο από όλε τι επιχειρήσει. Αλλά το 20% που είναι μεγάλο ποσοστό, 100 δι ευρώ. Αυτό το τμήμα λοιπόν σχετίζεται με μια ιδιαιτερότητα από χώρα σε χώρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα για να υπάρξει καλύτερη σχέση μεταξύ ευελιξίας από τη μία αλλά και ε, αυξημένης συγκρισιμότητας και να υπάρξει και ε, ελεγκτική σύγκληση. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες αρχές να μειωθεί για παράδειγμα και να μειωθεί η επίπτωση που θα έχει αυτό το στοιχείο στα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων και για το πώς θα προβλέψουν ε, τι απόδοση θα έχουν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού κάποια κριτήρια που βοηθούν μια ε, βελτίωση της αντικειμενικότητας αυτού του σημαντικού στοιχείου των ισολογισμών. Όλη αυτή η εργασία έγινε σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που μας βοήθησαν πολύ μέσω στοιχείων, μέσω συμμετοχής στην δημόσια διαβούλευση, μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τους ευχαριστώ θερμά όλους εφόσον ενδιαφέρονται τόσο πολύ να μας βοηθήσουν εμάς τις ΕΙΟΠΑ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να λειτουργήσει η φερεγγιότητα 2. Μια ευρύτερη αναθεώρηση θα γίνει λίγο αργότερα σε 2-3 χρόνια. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ματνέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω τις επικείμενες α, τροπολογίες στην κατοξιδότηση πράξη για τη φερεγγιότητα 2. Ποιο είναι το υπόβαθρο για να εξηγήσω τη λογική προσέγγιση της αναθεωρήσεως. Ό,τι η οδηγία Omnibus 2 συμφωνήθηκε το 2013, μεγάλα τμήματα του περιεχομένου της κατεξοδότηση πράξης ήδη είχαν προβλεφθεί, είχαν δοκιμαστεί ποσοτικά σε μελέτη ποσοτικοποιημένη, όμως κάποιοι ενδιαφερόμενοι κύκλοι επιθυμούσαν κάποιες τροποποίησεις κυρίως όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλουχικών απαιτήσεων πριν την θέση σε ισχύ της κατεξοδότησης πράξεως, ούτως ώστε να αποφύγουμε εκτοχιασμό της ε, εισαγωγής του φορεγιότητας Διού θέλαμε να κάνουμε αναθεώρηση των κεφαλουχικών απαιτήσεων μέχρι το τέλος του 2008 και αυτή η δέσμευση συμπεριλήφθη στην τελογική σκέψη 150 της κατεξουσιοδότησης συμπράξεως. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ασχολήθηκε με αρκετή και τα θέματα που σχετίζονται με τι επενδύσει σαν τμήμα ε, του προγράμματο για την ε, ε ενιαία κεφαλαγορά, κυρίω τι γίνεται με τα, μακροπρόθεσμα, τα, τα, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων, διαθωτικέ επενδύσει και πολύ σύντομα θα καθεσπίσουμε για τους επενδυτές και ασφαλιστές απαιτήσει με έναν απλό, τυποποιημένο ε, τρόπο, διαφανή τρόπο μέσω τροποποίηση ε, των κατεξουσιών πράξεων για την Φερεγγιότητα 2 θέλουμε αυτές τις τροποποίησεις της κατεξοδότητες πράξεων σύντομα να τις προτείνουμε πέρα από τις αλλαγές που ήδη έχουν λάβει η χώρα η αναθεώρηση του 2018 μας παρέχει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τεχνητά ζητήματα που εφήγησαν κατά τη διάρκεια του αιτήματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ευλήθη το 2015 για υποβολή συμβολών. Ζητήσαμε την ΑΙΟΠΑ να μα παράσχει συμβουλέ και να λάβει υπόψη του στόχου τη ε, ενιαία αγορά κεφαλαίων και εντοπίσαμε κάποιου τομεί που έπρεπε να γίνει αναλογικότητα, τεχνικέ ασυνέπειε ε, και εισηγημένου ε, τίτλους και το ιδιωτικό χρέο, όπω αναφέρθηκε και πριν λάβαμε την τελική έκθεση της ΑΙΟΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου με διεξοδική ανάλυση περίπου 25 στοιχείων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΙΟΠΑ για την δουλειά που έκανε, που ήταν απληρέστατη για την έκθεση. Η ζωή πληροφοριών της ΑΙΟΠΑ, η συνδρομή της είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ποιοτική. Εμείς ε, διοργανώσαμε μια δημόσια ακρόαση για την αναθεώρηση της, του, του ε, κανονισμού στις 27 Μαρτίου για τη του 2. Συμμετείχαν περίπου 300 ε, ε, σύνεδροι και αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο εγχείρημα που οδήγησε στην τροποποίηση της κατησότηση πράξης. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύουν προσεκτικά τις συμβουλές που μας έδωσε η ΟΠΑ. Με προσοχή αναλύσαμε και την αξιολόγηση αντικτύπου της ΑΙΟΠΑ και τι βλέπουμε ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι καλωσορίζουν εν γέννη τις τεχνικές βελτιώσεις που προτείνει η ΑΙΟΠΑ και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο τεχνικό έχουμε μια αρχική θετική άποψη για τα περισσότερα στοιχεία που περιέχεται στην αναφορά και στις συμβουλές που δίνει η ΕΟΠΑ με την επιφύλαξη βέβαια της τελικής απόψης που διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τούτου λεχθέντος βλέπουμε ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι εξέφρασαν επικρίσουν αφορά την ίδια πρωτοβουλία της ΑΙΟΠΑ, τις συμβουλές που παρήχε κατά πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια των δημοσίων διαβουλεύσεων και στην Ακρόση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάρτιο, κυρίως την πρόταση για τον κίνδυνο των επιτοκίων, είναι ένα επίμαχο θέμα αυτό, θα οδηγούσε σημαντική αύξηση όσον αφορά τις κεφαλοχικές απαιτήσει για τους ασφαλιστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν αμφισβητούμε το ότι αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και εδώ η ΑΙΟΠΑ έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετικώς προτάσεις. Θα ήταν ίσως προτιμητέο να επανεξεταστεί το ζήτημα του κινδύνου των επιτοκίων σαν τμήμα της αναθεωρήσεως της οδηγίας που θα πρέπει να λάβει χώρα κανονικά το 2020. Αυτή η αναθεώρηση θα είναι μια ευρύτερη αξιολόγηση του αντιχτύπου της αφαιρεγιότητας 2 σε μακροπρόθεσμες ασφαλιστικές δραστηριότητες και συνεπώς θα επιτρέψει πληρέστερη εικόνα για όλα τα θέματα συνετής διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείε και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών, η Συμβουλή όσον αφορά τα αξιόγραφα τα μη συγμένα οδηγεί σε καλύτερη αντίληψη των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιριών σε αυτούς τους τίτλους και όσον αφορά το μη βαθμολογημένο ε, ε, χρέος, θα πρέπει οι ιδιωτικές επενδύσεις να καλύπτονται όσον αφορά τη συνετή ε, διαχείριση, όπως και ε, τα διάφορα ομόλογα εταιριών. Αυτά τα δύο στοιχεία συνδυασμένα θα πρέπει να διευκολύνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να παράσχουν χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία σύμφωνα με τους στόχους του όλου προγράμματος. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θέλουμε τροπολογίε για τη καταξιοδότηση του καταξιοδότη κανονισμού η 2 τα μέτρα να, ε, να εφαρμοστούν φέτος. Ξεκίνησα τις αρχικές μου παρατηρήσεις εξηγώντα τους λόγους για το προγραμματισμό αναθεωρήσεως της καταξιοδότηση πράξεως του 2018 όμως όπως αναφέρει και ο Φάουστο αυτή η αναθεώρηση δεν είναι το τέλος του δρόμου η προβλέπει αναθεώρηση τη ίδια οδηγία που θα λάβει η χώρα το 2020 όπου περισσότερε θεμελιώδει αδηγίες για τη φερεγγιότητα 2 μπορεί να εξεταστούν ε, το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιώσιμη χρηματοδότηση ε, ήδη αναφέρει ότι κανόνε τη στη διαχείριση για τι βιώσιμε επενδύσει ίσω είναι ένα τομέα που πρέπει να εστιαστούμε για την αναθεώρηση του 2020. Θα ζητήσουμε από την ΕΟΠΑ να παράσχει συμβουλέ σχετικά με αυτό αργότερα, αυτό το έτος θα ζητήσουμε επίσημα και αναλύουμε και το θέμα των επενδύσεων σε τίτλους με την ευρία έννοια του όρου και για αυτό το σκοπό ξεκινάμε μια μελέτη για το τι γίνεται για τις επενδύσεις ευχαριστικών ταιριών και των συνταξιωτικών ε, ταμείων σε εισηγμένους και μη εισηγμένους τίτλους και τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το τέλος του τρέχοντος ε, έτους. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας και με τα χαράς να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικά τα σχόλια που κάνατε και καταλαβαίνω πως ε, πολύ σύντομα θα έχουμε τα κείμενα, δηλαδή όταν λέμε πολύ σύντομα, μάλλον πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά προτείνω να ξεκινήσουμε με την ομάδα των διαπραγματευτών. Ο πρώτος συνάδελφος δεν είναι εδώ, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ομάδα των σοσιαλιστών. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπερές. Εκτός αν κάποιος θέλει να μιλήσει εκ μέρους του έλκα. Αλλά νομίζω ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχα ήδη ενημερωθεί. Οπότε η κυρία Μπερές και μετά έχουμε και κάτι διάγει που όποιον θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Κλίντ, σας έχω σημειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε και από την ΑΙΟΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας άκουσα και τους δύο και βλέπω πως οι ασφαλιστές σας έχουν ήδη μιλήσει και τα επιχειρήματά τους έχουν ήδη εισακουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός με ε, τις τιμές αλλά η ερώτηση δική μου έχει να κάνει με το εξής ο κίνδυνος εκεί που βρίσκεται ανεξάρτητο με το αν είναι το 2020 ή το 2021. Μήπως θα έπρεπε εδώ να έχουμε κάποιο είδους αξιολόγηση για να δούμε οι διακυμάνσεις που θα μας οδηγήσουν και αν θα υπάρξει πρόβλημα για την βιωσιμότητα ή για την ε, ε, καλή κατάσταση των ασφαλιστικών ε, εταιριών. Επίσης, στην αναθεώρηση αυτή υπάρχουν δύο-τρία θέματα τα οποία επανέρχονται πολύ συχνά στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι καταρχήν το πώς θα μπορούσουμε να ε, μειώσουμε ε, τα shock actions στην ε, μακροπρόθεσμη διατήρηση χαρτοφυλακίου. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με την φερεγγιότητα 2, αλλά πιο πολύ με το αν θα ξανανοίξουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά είναι ένα θέμα ε, το οποίο μας ανησυχεί, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο θέλει να φτάσει η Κομισιόν. Είναι σημαντικό το θέμα και επίσης έχουμε και το ερώτημα ε, της, ε, ε, των ισολογισμών των ασφαλιστών και εκεί έχουμε πάρα πολλές διακυμάνσεις και διαπιστώνουμε έναν υψηλό βαθμό αστάθειας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς το θέμα αυτό σκοπεύει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έχω και άλλα τρία σημεία στα οποία θέλω να σταθώ. Μου έχουν θέσει το εξή θέμα. Ε, εξωτερικό εμπόδιο, Οι ασφαλιστές εκεί έχουν κάποιες ανησυχίες για τις, ε, ε, ε, για τις επιπτώσεις αυτής της εξισορρόπησης, οι οποίες βέβαια θα τους επηρεάσουν αρνητικά. Εκεί έχουμε ε, θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να λύσουμε μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, και ίσως μέσω της νομοθεσίας. Τώρα, ε, ε, κλάδος ασφάλειας ζωής ή μη. Εκεί έχουμε μία διαφοροποίηση. Θα λάβουμε υπόψη κάποιες νέες εκτιμήσεις ή όχι. Και το τελευταίο... και το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα τη χώρα την οποία προέρχομαι, ανεξάρτητα με το αν έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση ή όχι, η οχι συμμετοχή. δίνονται κάποιες εξαιρέσεις ε, στη δρέχουσα νομοθεσία, αλλά δεν καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ πεδίο, ε, δηλαδή δεν καλύπτουμε τις στρατηγικές συμμετοχές και κυρίως ε, στη βιομηχανία. Τέλος, και ίσως θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει από το σημείο αυτό, γιατί αν ακολουθήσουμε τις προσπάθειες που έχουμε κάνει στην ε, ε, ομάδα υψηλού επίπεδου και επειδή ε, ό,τι εξέταση του θέματος έχουμε κάνει μπορεί πάντα να ξανανοίξει, τι θα γίνει με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και πώς θα τρέξει το θέμα αυτό πάντα παράλληλα με τη φερικιότητα 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τα σχόλιά σας πολύ σχετικά. Ο κύριος Φόξ εκ μέρους της ECR. <coughs> Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ, ΑΕΟΠΑ, για την παρουσίαση που κάνατε και να σας πω πως αρκετοί από τους ε, εμπλεκόμενους σε αυτό το παιχνίδι ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί φοβούνται πως οι όροι που επιβάλλουμε είναι πολύ περιοριστικοί και ο σχεδιασμός του περιθωρίου ε, κινδύνου ε, ουσιαστικά οδηγεί στο αντί να χρηματοδοτούμε την πραγματική ε, οικονομία να τοποθετούμε γύρω στα 200 δις ευρώ ε, ως εξασφάλιση για τις απαιτήσεις κεφαλαίων. Τι σημαίνει αυτό, υπερβολικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν Πώς θέλετε εσείς, η ΑΕΟΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσετε <coughs> πως οι εμπλεκόμενοι ε, παρακολουθούν όχι μόνο τις εξελίξεις στο παιχνίδι, αλλά είναι και κομμάτι των υπολογισμών και των αποτιμήσεων που κάνουμε, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε ένα σχήμα το οποίο θα είναι υπερβολικά περιοριστικό και δεν θα αφήσει ε, περιθώριο ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Mm. Ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης. Είμαι σκιώδης για, τον, για την ΕΖΑ. Ε, άρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους νέους κανόνες για, το, για τα ΕΖΑΣ. Ναι. Λοιπόν, η νέα αυτή η Φερικαιότητα 2 άρχισε να ισχύει από το 16. Και όλοι θεωρούν ότι βελτιώθηκε έτσι ο έλεγχος ε, των δομών των ασφαλιστικών εταιριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά προβλεπόταν από την οδηγία και μια διαδικασία αναθεώρησης που θα έπρεπε να ασχοληθεί το 2018 με τις ε, κεφαλαιακές ε, απαιτήσεις και το 2020 θα έπρεπε να είναι μια πλήρης ε, αναθεώρηση για να ελέγξουμε επιτέλους εάν ε, αυτά που κάνουμε είναι σωστά. Αντίθετα με αυτή την προσέγγιση που ήταν σταδιακή, δηλαδή περιορισμένα μέτρα το 2018 και περισσότερα το 2020, τώρα στην πράξη λαμβάνονται μια σειρά από μέτρα που όπως είπε και ο Άσλι θα έχουν ε, τρομερή επίδραση, επίδραση στις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Μειώθηκαν κατά πολύ κάποιες ρυθμίσεις και έχουμε και τις συστάσεις της ΕΙΟΠΑ, όπως το είπε και η Περβάος, όπως είπε και η πρόσωπος της Κομισιόν, ότι πρέπει να, να αξιολογηθεί και το κίνδυνος από τα επιτόκια. Άρα θα πρέπει να αλλάξει κατά ένα τέταρτο η απέτηση φερικιότητας. Αυτό που μου είπαν εμένα είναι ότι ε, η ΕΙΟΠΑ πάει υπερβολικά μακριά. Ίσως με υποστήριξη και βοήθεια από την Κομισιόν. Γιατί αυτά δεν είναι απλώς ε, τεχνικές προσαρμογές. Εδώ είναι ουσιώδεις τροποποίησεις που έχουν τεράστιες επιπτώσεις και για τις κεφαλαικές απαιτήσει για τις επιχειρήσεις. Και όπως είπε και ο Άσλι, και επί της δυνατότητα των αγορών να χρηματοδοτήσουν. Και αυτό θέλουμε. Δηλαδή, βεβαίως έτσι θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ε, θέτουμε κινδύνο ένα από τους στόχους της ε, Ένωσης Χρηματαγορών και Κέφαλη Αγορών καλύτερα. Είναι τεράστιες επιπτώσεις, τεράστιες αλλαγές. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει ε, να λαμβάνονται μόνο από τους συνομοθέτες και όχι να αποφασίζονται μέσω κάτεξιοδότηση πράξεων μετά από σύσταση της ΑΙΟΠΑ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. ask to the colleagues of the ENF if they wish to take the floor. Someone all, Mr. Okay. Mr. Stoloyan. Ωραία, ο κύριος Στολογιάν. Όχι. Α, εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ την ΕΙΟΠΑ για τη δουλειά της, τις τεχνικές συμβουλές και την Επιτροπή για τα σχόλιά της και για την επιτελεστήσα και επιτελούμενη εργασία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Τώρα, το μη αξιολογηθέν χρέος. Καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που προτείνεται. Σε πολλά νομοθετήματα Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τους εξωτερικούς οργανισμούς ε, αξιολόγησης. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Μέσω εργασίας για να είναι επιτυχημένες οι μεθοδολογίες μας, να είναι πλήρως εφαρμόσιμες από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, χωρίς να υπονομεύουμε το υψηλό επίπεδο προληπτικής προστασίας που θέτει η φερεγγιότητα. Για τις στρατηγικές ε, επενδύσεις σε τίτλους πολύ καλό θέμα στα πλαίσια της ε, ΟΝΕ. Δηλαδή, απλώς πρέπει να υποβάλει εκθέσεις σε ΙΟΠΑ ή θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν εάν θα μπορούσε να παρέμβει για να μειωθούν τα κριτήρια αστάθειας για τον κίνδυνο από τα επιτόκια σημειώνω αυτά που είπε η Κομισιόν και πρέπει να πω ίσως θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί αυτό στην ευρύτερη αναθεώρηση του 2020 ούτως ώστε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών. Το ανέφερε και η κυρία Μπερέζα. Λοιπόν, να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για τη μελλοντική αναθεώρηση. Να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής και της ΕΙΟΠΑ. Τι έχει γίνει και τι εργασία έχει γίνει. Και ποια είναι αυτά τα θέματα. Η προσαρμογή λοιπόν ε, της αστάθειας από τη σελίδα 100 και 109 της έκθεσης ΕΙΟΠΑ. βλέπουμε ένα σενάριο με βάση το οποίο όσοι, όσες εθνικές αγορές αντιμετωπίζουν περισσότερη αστάθεια διαπιστώνουμε ότι επωφελούνται λιγότερο από τα μέτρα αυτά. Οπότε, το ερώτημά μου είναι σωστό αυτό το χαρτοφυλάκιο με τις ε, αρχές αναφοράς, με τις τιμές αναφοράς. Μήπως θα ήταν καλύτερα να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για να καταλάβουμε καλύτερα σε τι βοηθούν αυτές τις προσαρμογές. Αν δεν θέλουν άλλοι συνάδελφοι το λόγο, μήπω να μα ξαναπεί η ΕΙΟΠΑ και μετά η Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια για τις ερωτήσεις. Οι προσαρμογές για την αστάθεια. Αυτό που ανέφερε η κυρία Μπέρες και εσείς κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα τμήμα της εποπτείας του μέτρου ε, και του, της μελέτης αντιχτύπου. Δημοσιεύουμε κάθε χρόνο μια έκθεση. Κάθε χρόνο η έκθεση καλύπτει ευρύτερο πεδίο και περισσότερες λεπτομέρειες. Φέτος ε, θα έχουμε την τρίτη έκθεση και προσπαθούμε να αναλύσουμε περαιτέρω το θέμα και να δώσουμε στους ενδιαφερόμενους κύκλους και στους θεσμούς όλους, όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ένα θέμα που χρήζει προσοχής, είναι σαφές, όχι τώρα, δεν είμαστε έτοιμοι τώρα. Πρέπει να γίνει υπό το φως της θεμελιώδους αναθεωρήσεως που αναφέρθηκε στην αρχή. Οι στατικές επενδύσεις σε τίτλους και το θέμα του χρέους, το μη βαθμολογημένο, το μη το μη βαθμολογημένο είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε. Ε, δεν έχουμε κάποια πρόταση σχετικά, διότι η συζήτηση μεταξύ των υποπτικών φορέων ε, δεν μας άφησε να καταλήξουμε συγκεκριμένη πρόταση. Κάναμε τη δουλειά μας, αν επιτρέπετε να το πω αυτό, δώσαμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, όλα τα στοιχεία για την τωρινή χρήση και για τις δυσκολίες όσον αφορά την χρήση αυτού του στοιχείου. Τώρα για το μη βαθμολογημένο, βαθμονομημένο χρέος, μη εξελογημένο χρέος, συγγνώμη, ε, το εξετάζουμε το θέμα επί κάποιο χρονικό διάστημα. Προσπαθούμε πάντα να διαθέσουμε περισσότερο προσωπικό, να βοηθήσουμε τους ασφαλιστές, να μην, βαθίζονται, να μην βασίζονται πολύ στην εξωτερική πίστοση. Πολλά έγιναν δεν ξέρω όμως αν στο μέλλον θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το θέμα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, για την ώρα. Η συμβουλή που παρεσχέθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί καλή βάση και πιστεύω ότι θα μας επιτρέψει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα επιτρέψει αυτή η συζήτηση και τα πορίσματα να είναι αποτελεσματικότερες για τον κίνδυνο των επιτοκίων. Παραδεχόμαστε κι εμείς ότι είναι ένα θέμα, ευαίσθητο μάλιστα. Προτείνουμε σταδιακή εφαρμογή, αν υπάρξει κάποια εφαρμογή, διότι έχουμε επίγνωση του αποτελέσματος, προσμετρήσαμε τον αντίκτυπο. Δεν είναι ότι δεν λάβαμε υπόψη με κάθε σοβαρότητα το θέμα Έχουμε 28 εποπτικούς φορείς στην Ευρώπη και πιστεύουν αυτοί οι φορείς ότι αυτή η συμβουλή έπρεπε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι το αρνητικό επιτόκιο που είχαμε επί κάποιο χρονικό διάστημα έδειξε τα όρια της παρούσης προσεγγίσεως που στην περίπτωση αυτού του ε, υποσυνόλου του επιτοκίου δεν είναι αρκετά ε, αποτελεσματική προσέγγιση σε σχέση με την πραγματικότητα που διαπιστώθηκε. Έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις και υπάρχει δυνατότητα να περιμένουμε για την πλήρη αναθεωρήση των μέτρων. Πώς να το πω. Προτείνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι λογικό από πλευράς τεχνικής αλλά βέβαια οι θεσμοί θα κρίνουν κατά πόσο η πρότασή μας είναι καλή, κατά πόσο πρέπει να ληφθεί απόψη, υπόψη μεταγενέστερα στην αναθεώρηση της Φερεγγιότητας 2. Βιώσιμη χρηματοδότηση αναφέρθηκε. Προσβλέπουμε στην επεξεργασία του θέματος. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσπαθούμε να κατανοήσουμε πού και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ε, είναι σημαντικό θέμα. Το σχέδιο δράσης είναι αρκετά ευρύ, αλλά πιστεύουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε και τα συνταξιδοτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο για να βοηθήσουν. Είμαστε στην αρχή του εγχειρήματο. Για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα Ίσως εάν το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μας δώσουν και άλλους πόρους θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιώσιμης χρηματοδότησης. Θα ήθελα να ζητήσω κάτι τέτοιο με αυτή την ευκαιρία όσον αφορά τον κίνδυνο του κλίματος και κάποιο παρεμφερέ ζήτημα όπω αυτό που συζητούμε. Είναι πολύ τεχνικά ζητήματα και χρειάζεται η σωστή επεξεργασία χρειάζονται κάποιοι εμπειρογνώμονε και κάποια τεχνογνωσία δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς τη βοήθειά σας όσον αφορά τους ε, πόρους. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Ήδη ξεκινάμε τις προσπάθειες και θα το εξετάσουμε ενδελεχέστερα. Τι άλλο. Δεν βλέπω να έχει αναφερθεί κάτι άλλο. Α, για το περιθώριο του κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση Εξετάσαμε συνιστόσα του περιθωριού ε, του κινδύνου, που είναι το κόστος του κεφαλαίου. Εντατικές οι εργασίες μας, στο τέλος, καταλήξαμε με μία πρόταση. Να παραμείνει το παρόν επίπεδο. Δεν υπήρχαν στοιχεία για κάτι άλλο. Εξετάζουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα που είχαμε. Δεν είδαμε στοιχεία που να δείχνουν ότι πρέπει να προτείνουμε αναθεώρηση του παρόντος κόστου κεφαλαίου για το περιθώριο του κινδύνου, για το θέμα αυτό καθεαυτό, ε, αυτό δεν ανήκει σε αυτή την προσπάθεια, στο παρόν εγχείρημα, αφορά περισσότερο την θεμελιώδη αναθεώρηση της φερεγγιότητας 2, κάτι θα γίνει στο μέλλον. Δεν μπορώ για την ώρα να πω κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον αυτό θα έπρεπε να απευθυνθεί στα κράτη-μέλη για το θέμα των ε, πόρων. Ξέρετε πως εμείς είμαστε πάντα υπέρ της στήριξη των υποπτικών αρχών, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο εταίρος από την άλλη πλευρά του τραπεζιτού, λόγω τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, τα δικά σας σχόλια και τα σχόλια της κυρίας Μπερές, ε, του κυρίου Κλίντς και του κυρίου Φόξ επικεντρώνουν στην ανάγκη του να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όπως επίσης εξασφάλιση ε, του δημοσίου συμφέροντος. Και όλα αυτά βρίσκονται ίσως και στον πυρήνα της ε, πολιτικής που χαράσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα σε δύο στάδια. Καταρχήν, θέλουμε να ξεκινήσουμε με κάποια στοχευμένα θέματα μέσω κατεξουδότηση πράξεων και θέλουμε να αφήσουμε κάποια άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως είναι ευρύτερα, ε, ευρύτερα πολιτικά θέματα ή φιλοσοφικά ζητήματα για την αναθεώρηση που θα γίνει μετά το 2020. Και εδώ συνδέω με τα όσα είπε ο κύριος Κλίντς, δηλαδή ότι υπάρχουν ουσιαστικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει ο συνομοθέτης ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ε, συνομοθεσίας. Για να μπω και στα συγκεκριμένα σημεία ο κίνδυνος με τα επιτόκια, το είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια, γνωρίζουμε πως αποτελεί κομβικό θέμα και το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Παράλληλα όμως, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια, δεν έχουμε δει ε, ε, κάποια, ε, κάπως να διαταράσσεται η αγορά από το θέμα αυτό ε, και επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και οι κυκλικές ε, επιπτώσεις οπότε αν ε, βιαστούμε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα αναλάβουμε δράση τη σωστή στιγμή και ίσως ε, καταλληλότερη χρονική στιγμή είναι κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ε, το 2020. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε πως πιέζει το θέμα για να αντιμετωπιστεί ήδη από το 2018. Για ε, τις συμμετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο νομίζω ότι αυτό ισχύει και εδώ ε, για τις μη εισηγμένες ε, θα γίνει η εξέταση το 2018, αλλά αναγνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα με το μεταχικό κεφάλαιο, είτε είναι αυτό εισηγμένο είτε όχι, και θεωρούμε πως αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε ε, ευρύτερα. Είναι δύσκολο να γίνει μέσω κατεξοδότηση πράξεων και είναι δύσκολο μέσα από αυτές να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα με τις συμμετοχές και ε, τα μετοχικά κεφάλαια μέσω αυτών. Πιστεύω ότι μετά από την έρευνα που ζητήσαμε να γίνει φέτος, καλό θα ήταν να περιμένουμε τα αποτελέσματα που θα λάβουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς και μετά να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των στρατηγικών ε, επενδύσεων ε, όπου τα κριτήρια για να εντοπίζονται αυτές οι στρατηγικές συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά περιοριστικά μας εμποδίζουν από τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και νομίζω ότι οι επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να εξεταστούν και αυτές στα πλαίσια της αναθεώρησης που γίνεται το 2020. Τώρα, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το χρέος και το μη αξιολογημένο ή μη αποτιμημένο χρέος, νομίζω ότι η καλύτερη σύσταση είναι αυτή της ΕΟΠΑ, ότι δηλαδή θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά πριν προχωρήσουμε και να δούμε και το όριο του 5% την οροφή αυτή στις συνολικές συμμετοχές για να είμαστε σίγουροι πως καταρχήν χρειάζεται αυτή η οροφή και να είμαστε σίγουροι πως δεν υποσκάπτει τους στόχους μας. Δηλαδή, το να έχουμε περισσότερες ιδιωτικές συμμετοχές, επενδυτικές συμμετοχές στην Ευρώπη και να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για τέτοιου είδους επενδύσεις. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κρίνουμε ότι δεν θέλουμε πλέον να διατηρούμε το κατόφλι του 5%. Τώρα, βιώσιμη χρηματοδότηση. Θέλουμε αυτό να το δούμε στα πλαίσια της αναθεώρησης πράξεις θα απευθύνουμε μία πρόσκληση στην ΕΟΠΑ σύντομα και είναι πολύ πιθανό να συμπεριλάβουμε κάποιες διατάξεις της κατεξουδίωτηση πράξης ε, για τις ε, υποχρεώσεις αντισυμβαλόμενου και όλα αυτά στα πλαίσια της αναθεώρησης του 2020 θα ξαναεξεταστούν έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να συμμετέχουν και αυτές με ε, κρίσιμο τρόπο στην οικονομική βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Uh, Σας ευχαριστώ. Δεν έχω εδώ τον εισηγητή να σχολιάσει τα συμπεράσματα αυτά, οπότε προφανώς θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στο θέμα. Ακούσαμε όμω τι ευκρινήσει που μα έδωσε η ΑΕΟΠΑ και ακούσαμε και την προσέγγιση την οποία έχει σκοπό να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι όλα αυτά ήδη μας έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία. Έχουμε σημεία σύγκληση και υπάρχουν άλλα στοιχεία στα οποία πιστεύω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια διαλόγου και για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις αλλά και για την ε, αναθεώρηση που θα γίνει αργότερα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμπεράνουμε αυτά τα οποία μόλις, ε, αυτά, να συμπεράνουμε με τον τρόπο τον οποίο μόλις σας ε, περιέγραψα και να κλείσουμε το θέμα αυτό ευχαριστώντας την ΕΟΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών και μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.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

Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε μετά την ε, διακοπή το σημείο 5 τροπολόγηση του κανονισμού 904 κάθος 2010 μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας για θέματα ΦΠΑ. Πρόταση της Κομισιόν του περασμένου Νοεμβρίου. Νέοι κανόνε για συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών για να κατοβοληθούν οι απάτε του ΦΠΑ με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και το συντονισμό των ε, δράσεων, ε, κοινή έλεγχη και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου σε ενωσιακό επίπεδο. Για να υπάρξει μία νέα κατάσταση για το ΦΠΑ στα πλαίσια του σχεδίου δράση για το ΦΠΑ που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016. Ο Συγητή είναι ο κύριο Ζήλε. Υπέβαλε 25 τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση για να διασφαλίσει την κυριαρχία των κρατών μελών για φορολογικά θέματα και την προστασία των δεδομένων. Ο Συγητή δεν είναι εδώ. Θα τον αντικαταστήσει ο κύριο Λούνε από το ECR και έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ε, ζητάει ειλικρινά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί και με συγχωρείτε που και εγώ καθυστέρησα λιγάκι να μπω στην αίθουσα. Ο συγητή, ο κύριος Ζήλε Ρόμπερτς, συμφωνεί ότι η διαμεθοριακή απάτη του ΦΠΑ είναι μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο παρόν σύστημα φορολόγησης των εμπορικών συναλλαγών. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν οι φορολογικές αρχές την επιτάχυνση των συναλλαγών. Η Κομισιόν παρουσιάζει σαφή στοιχεία. Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ συντελεστών ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών, αλλά είναι ακόμη 12,8 το 2015. 12,8 μονάδες, ποσοστίες μονάδες. Και μεταξύ ορισμένων κρατών μελών ε, υπάρχουν διαφορές και άνω του 20%. Των 20 ε, ποσοστίων μονάδων. Όλα αυτά δεν είναι θέμα Βεβαίω ε, απάτης, αλλά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι τμήμα. Είναι τμήμα για τη διαφορά στην συλλογή του ΦΠΑ μεταξύ κρατών μελών. Ο συγητής καλωσορίζει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, για να καταπολεμηθεί η απάτη του ΦΠΑ ταχύτερα, ευκολότερα, πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, αν εξετάσετε την πρόταση, ο εισηγητής έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές που θεώρησε αναγκαίες. Γιατί θεωρεί ότι η πρόταση αυτή πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ από τη μία πλευρά τα αιτήματα για αποστολή πληροφοριών και την ανάλυση τους και από την άλλη πλευρά την προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Γι' αυτό έχουν προταθεί τροπολογίες για να οριστούν τα επιχειρησιακά όρια του Eurofisk και η επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών από διάφορες αρχές. Γίνονται αναφορές σε διάφορα νομοθετήματα για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, η πρόταση βελτιώνεται για να υπάρξει καλύτερη λοιπόν ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των ε, ευθυνών των αρχών που ζητούν και των αρχών που λαμβάνουν πληροφόρηση χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα να ξεκινήσουν διοικητικές έρευνες οι αρχές που ζητούν πληροφόρηση και να λάβουν καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης προβλέπεται απλουστευμένος μηχανισμός για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις, ε, ε, ε, τα χρέη ΦΠΑ τα κράτη-μέλη. Οι τροπολογίες επίσης στοχεύουν στην διευκρίνηση και τη σαφήνεια του κειμένου και του πνεύματος της οδηγίας. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την παρουσίαση από πλευρά του συγητή. Ισκιώδης τώρα. Τρία λεπτά παρακαλώ καθένας, αλλά θα είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι. Καμπριέλ Μάτο, Έλκα. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόμπερτς για την πρότασή του την οποία θεωρώ θετική. Με την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς όχι μόνο είναι επιθυμητή αλλά απόλυτα αναγκαία η συνεργασία των αρχών των διαφόρων χωρών. Το καθεστώς ΦΠΑ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στο ρυθμό της παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης. Οπότε οι προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας είναι ακόμη πιο χρήσιμες. Χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση για να καταπολεμηθούν οι απάτες και για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά. Αλλά θέλω να είναι σαφές ότι περισσότερη εναρμόνιση δεν σημαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Σημαίνει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Καλή συνεργασία για να γίνεται σωστός έλεγχος. Η Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης για τον ΦΠΑ τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ΦΠΑ για να εμπλουτιστούν οι προκλήσεις του παρόντος αιώνος και μέσω πρόθεσμα θα προτείνει μια σειρά ουσιώδη μέτρα για να εξυγχρονιστεί το σύστημα του ΦΠΑ, να απλουστευτεί και να γίνει πολύ πιο ανθεκτικό στην αντιμετώπιση των απατών και πιο επιβοηθητικό των επιχειρήσεων γιατί αυτό το σημερινό βήμα εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που θέλω να τονίσω αφορά πρώτα απ' όλα το άρθρο 7. Πρέπει όταν ε, ζητείτε από κάποιο κράτος μέλος από άλλο μία δυτική έρευνα, διοικητική έρευνα πρέπει να διεξάγεται δεν θα είναι δυνατόν αυτός που λαμβάνει το αίτημα να αρνηθεί την εκπλήρωσή του. Είναι θεμελιώδες. Εφόσον υποβάλλεται το αίτημα, πρέπει να εκτελεστεί, γιατί αλλιώς το κράτος μέλος το οποίο ζητάει κάτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα εφόσον ε, το υποκείμενο του αιτήματο είναι σε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει λοιπόν να καθοριστεί σωστά ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι υπάλληλοι του ετούντος ε, κράτους στις διαδικασίες ε, του κράτους που θα πρέπει να εκτελέσει το αίτημα. Επίσης, η παρουσία υπαλλήλων στην, ε, στις υπηρεσίες του άλλου κράτους και στα γραφεία και καταστάσεις του υποκειμένου της έρευνας. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να το επιβάλλουμε. Και μια άλλη καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στο 10ο κεφάλαιο. Η δημιουργία του Eurofisk για να διευκολυνθεί η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί η απάτη μεγάλης κλίμακας ή οι νέες μέθοδοι απάτης στον ΦΠΑ. Πρέπει λοιπόν Δεν πρόκειται βεβαίως να αφαιρέσουμε εθνικές αρμοδιότητες ε, για τη φορολογία των κρατών μελών, αλλά χρειάζεται στενή συνεργασία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα για να επιτύχουμε τους στόχους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουμε να συνεργαζόμεθα και παραλαμβάνω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή και σε εσά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ο κ. Λούντβιξον, που είναι σκιώδης για τους S&D, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, για αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σειρά μέτρων που αφορούν το ΦΠΑ και πιστεύω ότι είναι θεμελιώδου σημασία το έργο πραγματοποιούμε να είναι αποτελεσματικό. Να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη όσον αφορά το ΦΠΑ. Είναι ε, φορολογική απάτη, απάτη του ΦΠΑ. Η πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έκανε τις 13 Νοεμβρίου του 2017 ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Ο εισηγητής αναφέρεται στην προστασία των στοιχείων, των δεδομένων και την ακαιρεότητα των προσώπων. Εν γέννη προβλέπεται ε, προστασία ε, των δεδομένων και πρέπει να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να γίνει πιο εντατική δουλειά για την καταπολέμηση της ε, απάτης και της φοροδιαφυγής και κυρίως της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργοποιηθούν σε αυτό το τομέα, να ενισχυθούν σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών όσον αφορά υπόνοιες απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Πρέπει να βελτιωθεί αυτός ο τομέας. Ε, οι διάφορες φορολογικές αρχές θα πρέπει να επομιστούν τις ευθύνες τους όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου και θα πρέπει να κινηθούν επικοδομητικά θα πρέπει να βοηθούν τις διοικητικές έρευνες που διενεργούνται για την καταπολέμηση των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις φορολογικές αρχές του το τρόπος. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής αναφέρεται σε πιστοποίηση, αλλά θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασίας, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε στέρεα ισχυρά φορολογικά συστήματα και αυτό θα επιτρέψει να θεωρείται αυτός που υπόκειται στην υποχρέωση του ΦΠΑ σαν φορολογούμενος εν γέννη. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που μπορούμε να το συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε εντατικά για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις θα πρέπει να επιτεθούμε κατά των εγκληματικών ομάδων που κάθε χρόνο διαπράττουν πολύ σημαντικές απάτες στο ΦΠΑ και αυτό αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια ευρώ απώλειες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν έχουμε αποκλίνηση απόψε κάποια σημεία τελικά θα καταλήξουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον εκπρόσωπο της Άλντε που θέλει να λάβει το λόγο, ούτε για την ΚΟΕ αλλά οι πράσινοι θέλω να λάβουν το λόγο. Η εκπρόσωπο των πρασίνων, ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Λούτβικσον και εμεί υποστηρίζουμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία και θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο, να ενισχύσουμε τη συνεργασία των κατώμελων για την καταπολέμηση των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το σχέδιο εκθέσεώς του, αλλά έχουμε κάπως διαφορετική άποψη από αυτού και θα υποβάλουμε διάφορες σχετικές τροπολογίες. Είδαμε τις τροπολογίες του που αφορούν την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τροπολογίες του δεν μας βρίσκουν απολύτω συμφώνους. Δεν είμαστε υπέρ διαγραφή της αναφοράς στην έννοια των πιστοποιημένων φορολογουμένων ατόμων ε, είναι ε, μια ιδέα που αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να εξετάσουμε αυτή την έννοια του φορολογούμενου στον τομέα του ΦΠΑ και μπορούμε να αλλάξουμε την έννοια αυτή, αλλά δεν θέλουμε διαγραφή, όπω προτείνει ο συγγετή. Συμπελέμβανε και τροπολογία στου συγκεκριτή για την προστασία των δεδομένων και φοβούμεθα ότι αυτό ίσω να είναι κάτι πολύ περιοριστικό όσον αφορά τι αναγκαίε ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά τα φορολογικά μεταξύ κρατών μελών. Βεβαίω, υποστηρίζουμε πλήρω την ανάγκη για την προστασία των δεδομένων και ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά δεν θα θέλαμε συμπεριθεί στο κείμενο διότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τα κράτη-μέλη σαν ένα τρόπο μειώσεω τη συνεργασία του όσον αφορά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Κατάλληλο ηγητή τροποποίησε μια τη βασικέ διατάξει προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι η ετούσα αρχή θα πρέπει να έχει την ίδια δυνατότητα ελέγχου που έχει το κράτο προ η αίτηση. Λοιπόν, η αναφορά τη εξουσία έρευνα δεν αναφέρεται στο κείμενο και είναι βασικό στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά η συνεργασία. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι τα μέσα για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση τη απάτη του τομέα ΦΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε μέσα των τροπολογιών μα. Καταρχά, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα κοινών ελέγχων που πιστεύουμε ότι είναι μια βελτίωση σε σχέση με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι κάτι που ζητήσαμε κατά το παρελθόν θα επιδιώξουμε την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και συνεργασία με την Europol, Eurofisc και την OLAF και με το PPO, με το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για τις πιο σοβαρές υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και δεν θα πρέπει να υπάρχουν νομικά ή διοικητικά εμπόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών για να βελτιστοποιηθεί η προσπάθεια ε, καταπολέμησης των παρανόμων οργανώσεων. Και τέλος θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ρήτρα για τα πλέον ευνοούμενα κράτη εντός του κανονισμού του ΦΠΑ για τη διοικητική συνεργασία κάτι παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στο ίδιο το ΝΤΑΚ για την άμεση φορολόγηση, ούτω ώστε όταν η αρμόδια αρχή ενό κατου μέλου παραλάβει κάποιε πληροφορίε από τρίτη χώρα, αυτή η αρχή έχει τη δυνατότητα να διαβάσει πληροφορίε στα κράτη-μέλη τα οποία σα ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με του κοιόδη ηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι σκιώδει. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλουν να λάβουν το λόγο. Και μετά κάτσε και θα το κλείσουμε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που στήριξαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το είπατε κι εσείς, είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο στην προσπάθεια αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ και θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε επιπλέον εργαλεία έτσι ώστε υπό το τρέχον καθεστώς να καταπολεμήσουμε την ε, ε, αποφυγή ε, πληρωμής ΦΠΑ και τα θέματα τα οποία θέσατε εσείς είναι όντως τα πιο σημαντικά της πρότασης. Αυτή τη στιγμή γίνονται εντατικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Συμβουλίου, αποτελεί προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας και να συμπληρώσω πως η μεγάλη καινοτομία αυτού του κανονισμού είναι η δυνατότητα υποχρεωτικής διοικητικής ε, έρευνας και κυρίως όταν δύο κράτη-μέλη ζητήσουν από ένα τρίτο να κάνει κάποιο είδους ε, έρευνα. Αυτή είναι μια καινοτομία γιατί επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να ελέγχουν ε, τις συναλλαγές που γίνονται στα πλαίσια του νέου ε, νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο που πολύ σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα για τη διαγραφή των διατάξεων για τα θέματα CTP να σας πω ότι συμφωνήσαμε με τα όσα μόλις ακούστηκαν και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άδρα αυτά εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι. Δεν θα την αποσύρουμε. Παράλληλα όμως δεν θα πρέπει ε, να παρακολουθήσουμε τη συμφωνία για τα υπόλοιπα κομμάτια ε, του κανονισμού. Η πρόταση, επαναλαμβάνω, παραμένει στο τραπέζι, θα τη διαπραγματευτούμε και θα τη διαπραγματευτούμε γενικότερα κάποια από αυτά τα θέματα στα πλαίσια της αναθεώρησης του καθεστώτος ΦΠΑ. Τώρα, συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών, Όλαφ Europol και εδώ θεωρούμε πως προσφέρουμε μια ε, μεγάλη καινοτομία ε, μέσα από το κείμενο αυτό και ότι δεν θα πρέπει οι πληροφορίες που μπορούν να τύχουν ε, ανταλλαγής να μην περιοριστούν υπερβολικά. Είναι όντως ευαίσθητο το θέμα για κάποια κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να βρούμε μια εύχρηστη λύση που να μας εξυπηρετεί. Προστασία δεδομένων, τέλος. Έχετε δει τις προτάσεις μας σχετικά όπου ενημερώνουμε τις διατάξεις έτσι ώστε να ε, ευθυγραμμιστούμε με τις πιο πρόσφατες ε, τροποποιήσεις και πιστεύω πως θα πρέπει να ε, ενημερώσουμε έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε το στόχο μας. Δηλαδή όχι να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη από το να συνεργάζονται αλλά να εξασφαλίσουμε πως τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται χωρίς όμως αυτό να παρεμποδίζει από τη συνεργασία και την ανταλλαγή. Ουσιαστικά δηλαδή θέλουμε ένα κείμενο το οποίο στο σημείο αυτό να έχει ισορροπία. Περνάμε στο Catch the λοιπόν μετά από εσά και είδα πως πρώτη έχει ζητήσει το λόγο κυρία Μπερέσου. Ευχαριστώ. Κοίταξα με πολύ προσοχή τις ε, προτάσεις ε, του εισηγητή και ευχαριστώ αυτόν και τους υπόλοιπους ε, ομιλητές. Τώρα, να συμπληρώσω στα όσα είπε ο Σκιώδης κύριος Λούτφίξον, γιατί συμφωνώ με όλη την ανάλυση που έκανε, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ. Τι διακυβεύεται μέσω της πρότασης αυτής. Διανύουμε μία στιγμή όπου σε επίπεδο διοικητικής συνεργασίας έχουμε προχωρήσει πολύ. Και εδώ θα προχωρήσουμε και στο χώρο του ΦΠΑ. Και έχω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα μιας πολύ ωραίας συνεργασίας ε, διοικητικής ε, της συμφωνίας που συνάψαμε πρόσφατα με την Ορβηγία. Και νομίζω πως είναι ένα κείμενο το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήταν λοιπόν παράξενο για τη διοικητική συνεργασία με την Ορβηγία να έχουμε μια υποδειγματική συμφωνία, φιλόδοξη, και να μην τη χρησιμοποιήσουμε ως μοντέλο ή μέτρο σύγκρισης για τα όσα θα κάνουμε σε επίπεδο διοικητικής συνεργασίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί διαβάζοντας κάποιες από τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας και που έχει καταθέσει ο εισηγητής, θεωρώ ότι απομακρυνόμαστε από αυτό το μοντέλο και θα έπρεπε τουλάχιστον σε επίπεδο φιλοδοξίας να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα πετύχαμε εκεί. και θα πρέπει να εμπνευστούμε από το πνεύμα το οποίο διέπει όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για τη διοικητική συνεργασία ε, στην ΤΑΚ και ίσως ε, και σε άλλα πεδία εκτός από το πεδίο του ΦΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κανένα συνάδελφο. Θα ζητήσω λοιπόν από τον εισηγητή να κάνει κάποια σχόλια. Α, εσείς τον εκπροσωπείτε μάλιστα. Όχι, δεν έχω κάτι ακόμα. Ε, περιμένει με χαρά να συνεργαστεί και στα υπόλοιπα σημεία. Λοιπόν, 23 Μαΐου, 5 το απόγευμα, τροπολογίες. 18 Ιουνίου θα συζητηθούν. 19 Ιουνίου ψηφίζουμε στην ΕΚΟΝ. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Θα διακόψουμε τώρα για 7 λεπτά για να περιμένουμε τον κύριο Φάρμπερ που είναι ο εισηγητής των επόμενων δύο θεμάτων. Επτά λεπτά διάλειμμα και τα ξαναλέμε.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 Uh, Ευχαριστώ πολύ Μάρκους. Διαφορετικ... Υπάρχουν διαφορετικέ ε, απόψει τα χρονοδιαγράμματα λόγω διαφορετικών προεδριών που έχουν διαφορετικέ απόψει. Θα επιληθεί. Θα επιληθεί το θέμα. Μίλησα με του Βούλγαρου και του Αυστριακού. Δεν ξέρω αν υπάρξει και άλλη Αυστριακή Προεδρία. Θα δούμε, το ρυθμίσει η Γραμματεία. Ελπίζω να είναι δικαιολογημένη η αισιοδοξία σα για τους σοσιαλιστές. Η Περβάνς αντικαθιστά τον Σκιώδη. Ευχαριστώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ένα σημείο που πρέπει να διαβάσω εκπροσωπώντα το σκιώδη μα, αλλά έχω και τη δική μου άποψη θέλω να εκφράσω. Ίσως πρόεδρε αν επιτρέπετε θα προσπαθήσω να συνδυάσω και τα δύο σκιοδησηγητής, ε, η κυρία Ντελβό ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα. Είχε σημαντική συνεδρίαση στο Παρίσι. Οπότε θα διαβάσω την άποψή της. Καλωσορίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύει ότι είναι καλή. Θα βοηθήσει θα ενισχύσει το καθεστώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδυτικές θα βγουν από το τραπεζικό πλαίσιο το CRR και το CRD και αυτό συνάδει με το στόχο να αποφευθούν κενά όσον αφορά τη λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Είναι μια πρόταση για προληπτικές απαιτήσει που προσαρμόζονται καλύτερα στο, στους διάφορες μορφές κινδύνου, στο διαφορετικό μέγεθος των επιχειρήσεων, διότι επενδυτικέ εταιρείε δεν έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικά και λιανικής. Ταυτόχρονα διορθώνονται κάποιες καταστάσεις όπου κάποιες εταιρείε έτυχαν εξαιρέσεως και δεν υπόκεινται σε απαιτήσει προληπτικής ε, προσέγγισης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις. Εκτιμά και την απλή και σαφή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως πιστεύει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η απλότητα δεν αντιβαίνει του στόχου μας να έχουμε ισχυρό πλαίσιο για την αγορά αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επενδύσεις που χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό καλωσορίζει την προσέγγιση του κυρίου Φερμπερ για μεγαλύτερη αναλογικότητα και θέλει να τον ευχαριστήσει για την έκθεσή του. Ε, εντόπισε, εντυπωστήκαν 11 διαφορετικά είδη επενδυτικών επιχειρήσεων το να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες όλες αυτές οι εταιρείες είναι κάτι πολύ δύσκολο και πιστεύει ότι θα υποβάλει σχετικέ τροπολογίες για να ρυθμιστεί κατάλληλα η πρόταση ούτω, ώστε να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες για τα διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα και για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Δεν είναι σίγουρη για το ποια προσέγγιση δίνει στις αρμόδιες αρχές μεγάλη διοικητική ευχαίρεια ε, και δεν ξέρει αν η νομοθεσία του δευτέρου επίπεδου εγγυάται την αλογικότητα. Αναφέρει ότι οι επενδυτικές εταιρείες, 80% ε, ε, αυτών βρίσκονται στον Αμένο Βασίλειο και αυτό σημαίνει ότι αυτό το χαρτοφυλάκι έχει διάσταση Brexit. Οπότε καλωσορίζει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στοιχεία, για ισοδυναμία. Είναι κάτι ισορροπημένο που κινεί προ σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, συνεχιζόμενε διαπραγματεύσει για την έκθεση για την ισοδυναμία είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη και εδώ και πέραν αυτού πιστεύει ότι το θέμα των κανόνων περί συνδυάζεται με την ολοκλήρωση των τεσσάρων θεμάτων του CRD διότι υπάρχουν διάφορες μορφές κινδύνου ε, ε, όσον αφορά την αναλογικότητα. Πρέπει αυτέ οι εταιρείε να έχουν ε, πιο ήπια αντιμετώπιση από ό,τι τράπεζε και χρειάζεται το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα να έχουμε μια αναβολή για τουλάχιστον ένα μήνα για αυτά τα θέματα. Και ας συντονίστρια του S&D πρέπει να πω ότι ένθερμα υποστηρίζω αυτό το αίτημα αλλά Πρόεδρε το θέμα είναι θέλετε να προσθέσω την πρότασή μου στα πλαίσια του Catch the Eye ή να δευτερολογήσω μετά. Παρακαλώ σημειώστε με στον κατάλογο το ώστε να ξαναπάρω το λόγο αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τις ομιλίες των σκιωδών θα λάβετε το λόγο. Κύριος Λούκε από το ECR. Ευχαριστώ. Θεμελωδώς θεωρώ ότι είναι καλή προσέγγιση της Κομισιόν δημιουργούνται αυτές οι τρεις κατηγορίες ε, εταιρεών επενδύσεων. Είναι λοιπόν μια ταξινόμηση όσον αφορά τις ε, προληπτικές προϋποθέσεις ε, κεφαλαιακής επάρκειας. Συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Φέρμπερ ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει προσαρμοστεί κυρίως ε, στον τρόπο με τον οποίο ε, ελέγχονται οι τράπεζες. Οπότε, όταν θέλουμε να μειώσουμε το ρυθμιστικό άχθος, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Να διακόψω μέχρι να μπορείτε να με ακούσετε. Υπάρχουν δύο λοιπόν δυνατότητες έλεγα. Είτε να πούμε θέλουμε κυρίως να ε, διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των ε, χρηματαγορών ή κυρίως θέλουμε να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός με τις τράπεζες που επίσης ε, συμμετέχουν σε αυτές τις χρηματαγορές. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επιλέξουμε την πρώτη λύση. Δεν θα πρέπει οι απαιτήσει έναντι αυτών των εταιριών να μην βοηθούν τη σταθερότητα των αγορών αξιογράφων. Έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο λειτουργίας αυτές οι εταιρείες. Ορισμένες είναι απλώς ε, εταιρείε προσωπικέ. Πρέπει να μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ. Γι' αυτό υπέβαλα τροπολογίε. για να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής και θεωρώ ότι ο ΕΣΜΑ πρέπει να ε, έχει περισσότερο κύρος έναντι της EBA γιατί μέχρι στιγμής κυρίως η EBA παίζει τον πρώτο ρόλο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή τη δυναμική. Δεύτερον, ποιες είναι οι, πραγματικά οι μικρές εταιρείε που δεν είναι εισηγμένε. Νομίζω ότι είναι αυστηροί οι περιορισμοί που τίθενται. Για ορισμένους τομεί δραστηριότητας ε, λένε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει καμία δραστηριότητα, μηδέν. νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε κάποιες ε, λειτουργίες και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε φραγμούς για νέες εταιρείε που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις αγορές. Επίσης, δεν νομίζω ότι μια τέτοια νομοθετική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει και τον τρόπο καθορισμού των αποδοχών ή υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Εάν οι εταιρείε δεν έχουν καμία συστημική σημασία, δεν πρέπει να τους ε, υπαγορεύουμε να δημοσιοποιούν ε, το καθορισμό των αποδοχών για τις ε, συνθήκες για τις εταιρείε από τρίτες χώρες Συμφωνώ με τον κύριο Φάρμπερ, η ισοδυναμία είναι ο καλύτερος τρόπος. Πρέπει να, υπάρξει, πρέπει να, υπάρχει, να υπάρξουν ανοιχτές αγορές, να βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό. Οπότε κύριε Φέρμπερ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την τροπολογία μας 28. Μήπως μπορείτε στις καταληκτικές παρατηρήσεις να την εξηγήσετε. Αλλά αν θέλουμε να μην επιτρέπουμε αυτά που προβλέπει το MIFID για τις εταιρείε τρίτων χωρών, τότε θα τις υποχρεώσουμε να αλλάξουν έδρα. Νομίζω ότι είναι φραγμό στον ανταγωνισμό στην ουσία είναι προστατευτικό μέτρο. Άρα δεν βοηθάμε τον ανταγωνισμό, δεν βοηθάμε το άνοιγμα των ε, κεφαλαίων αγορών. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον από τους φιλελεύθερους. Δεν βλέπω κάποιον. Ο κύριος Λάμπερτς για τους πράσινους, αλλά νομίζω κάποιος θα τον αντικαταστήσει. Και ο κύριος Γκυγκόλ είναι επόμενος. Δεν είμαι από την ΚΟΕ, είμαι πάρα πολύ υπέρ της Ευρώπης και μη λέτε ότι είμαι από την ΚΟΕ, δεν έχω σκοπό να μετακινηθώ, θέλω καταρχήν αυτό να το επαναλάβω. Και δεν ξέρω γιατί είστε εσείς στην ΚΟΕ. Ξέρω πως οι σοσιαλιστές προσπάθησαν να σας προσελκύσουν και ξέρω πως απέτυχαν. Εν πάση περιπτώσει, πρόεδρε, μου έχετε δώσει το λόγο ή όχι. Uh, ναι, ε, ε, σας είχαμε σημειώσει λάθος στα έγγραφα, ας το αφήσουμε εκεί και σας δίνουμε το λόγο. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πρόταση η οποία σε γενικές γραμμές είναι καλοδεχούμενη. Και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για ένα μεγάλο κομμάτι των τροπολογιών του και πρέπει να σου πω ότι με χαρά περιμένω να γίνει και η συζήτηση. Οι πράσινοι πάντα συμφωνούσαν στην αναλογικότητα στους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και πώς οι κανόνες θα πρέπει να βασίζονται σε μια πραγματική ανάλυση του ποιοι κανόνες είναι απαραίτητοι για ποιο επιχειρηματικό μοντέλο. Κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τον εισηγητή και πιο συγκεκριμένα αυτές που σχετίζονται με τα παραθυράκια ε, για τα SI είναι πολύ καλές γιατί κλείνουν τα παραθυράκια εκεί και μάλιστα οικοδημούν ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε αξιολόγηση ε, διαδοχικών ετών ε, και εξασφαλίζουν ε, ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλα τα κράτη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε. Uh, Κοιτώντα τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακούγοντα ανησυχίε και των πολιτών και πολλών συμμετεχόντων, είναι οι κατηγορίε. Οι κατηγορίε που δημιουργήθηκαν βασίστηκαν στα σωστά κριτήρια. Γιατί αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι αφενός μέχρι στιγμής έχουμε ένα υπερβολικά περίπλοκο ε, σύστημα για τους μικρότερους και όχι τόσο σημαντικούς παίκτες και μετά για τη διαχείριση αφιερώνται τεράστια ποσά. Ε, τα κεφάλαια δεν πρόκειται να ενισχυθούν με ισχυρότερους κανόνες, δεν πρόκειται ε, να τους παρακολουθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρόλο που μερίδιο αγοράς μπορεί αυτές οι εταιρείε να έχουν τεράστιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια είναι η δύναμη η εξουσία που έχουν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού ε, σε αυτό το σενάριο. Και τα κριτήρια τα οποία αυτή τη στιγμή βασίζονται μόνο σε αριθμητικά στοιχεία και σε ίδια κεφάλαια θα πρέπει να λάβουν υπόψη στους υπολογισμούς τους και ποιοτικά στοιχεία, για παράδειγμα, το πώς επηρεάζουν ε, μία ε, αγορά ε, κοινωνικής οικονομίας. Δεν θα έπρεπε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί νομίζω ότι πολλές οι επιχειρήσεις είναι ε, αυτές οι οποίες ζητάνε να έρθουν σε επαφή μαζί μας γιατί θέλουν να αντιμετωπίσουν την υπερβολική ισχύ αυτών των ε, διαχειριστών ε, κεφαλαίων που περιγράφονται εδώ. Μήπως λοιπόν στον υπολογισμό των κεφαλαϊκών απαιτήσεων θα πρέπει να συμπληρώσουμε με κάποια κριτήρια ακόμα. να το σκεφτούμε πιο προσεκτικά γιατί μπορεί κανείς για παράδειγμα να μηνυθεί ε, και αν δεν έχει επαρκή κεφάλαια το δικαίωμα αποζημίωσης ε, χάνεται. Βλέπω βέβαια ότι ε, εξαρτάται από το αν οι επιχειρηματικές αυτές συμβουλές είναι discretionary ή όχι, αλλά το σύστημα το οποίο δημιουργείται είναι υπερβολικά περίπλοκο και πρέπει να σας πω πως σε όλη την γάμα κάνουμε κάποιου είδους ε, καινούργιες εισαγωγές με κινδύνους, οι οποίοι είναι κοινωνικοί, είναι περιβαλλοντολογικοί, είναι εταιρικοί και δεν είναι αρκετά διάφανοι. Και θα ήθελα μέχρι τα τέλη του μήνα να έχουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να καταθέσουμε τροπολογίες οι οποίες θα λάβουν υπόψη και τα στοιχεία αυτά για τις επενδυτικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα όπως πρέπει. Τέλος, πιστεύουμε πως εκ των προτέρων κάποιοι κανόνες και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Λούκε εκ των προτέρων κάποιοι κανόνες θα πρέπει να είναι ανακράτος ε, και στην υποβολή φορολογικών ε, στοιχείων αλλά και για κάποιου και για συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα να εισαχθούν γιατί αντιμετωπίζουμε τον εξής κίνδυνο. Εμείς να μην δούμε ε, κινδύνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή υφίστανται. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση και πιστεύω πως η αναλογικότητα η οποία έχει εισαχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ιδέα της απλοποίησης θα πρέπει να συνοδευτούν από ισχυρότερους, στεναρότερους κανόνες για αυτούς που είναι οι πιο δυναμικοί παίκτες στην αγορά, που σε μία ε, ε, οικονομία κοινωνικής αγοράς ενισχύονται συνέχεια και οι οποίοι δεν υπήρχαν όταν δημιουργήσαμε εμείς την ενιαία αγορά στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω τώρα ε, να είναι σωστά οι, σωστά οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν αναγραφεί. Ο κύριος Βιάγκας δεν είναι εδώ, οπότε ποιος είναι από την ΚΟΕ. την Επιτροπή μας ότι δεν είναι εδώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ε, και είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες θα συμβάλλει με παρατηρήσεις και τροπολογίες. Δεν ήθελα να τον αντικαταστήσω. Απλώς ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Γκίγκολτ. Ε, θα μπορούσε να διορθώσει το λάθος σας, γιατί τον αναφέρατε ως εκπρόσωπο της Ευρωμάδας της Αριστεράς, αλλά θα τον παρακαλούσα να σέβεται περισσότερο και την Ευρωμάδα της Αριστεράς και εμένα προσωπικά αυτά που είπε για την Ευρώπη και τα λοιπά ως σχόλια και για τους σοσιαλιστές τα θεωρώ και ατυχή και άδικα και επειδή είναι καλός συνάδελφος και φίλος θα ήθελα δημόσια εδώ στη συνεδρίαση να τον παρακαλέσω να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα. Thank you. I guess you can, you can... Ευχαριστώ. Μπορεί να το λύσετε εκτός της αίθουσας αυτό το θέμα προτείνω να πάμε στη δικασία Catch the Eye και μετά θα ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο, μετά στον εισηγητή ο λόγος και μετά θα ολοκληρώσουμε. Για η κυρία Σάντερς και η κυρία Μπέρε είναι οι πρώτοι που θα πάρουν το λόγο. Στο Eye. ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις που έκανε και θα ήθελα να προβώ σε ένα σχόλιο όσον αφορά τις διάφορες διατάξεις που αφορούν τι τρίτες χώρε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις εν λόγω διατάξεις, οι ιδιαίτερος να ενισχύσουμε αυτή που υπάρχει στο ΜΙΦΙΡ. Αυτοί οι κανόνες ε, δεν είναι πάντα απόλυτα σαφείς, ε, δεν είναι πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και η ισοδυναμία που υφίσταται δεν επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο είδη προβλημάτων κατά την άποψή μου. Το πρώτο είναι όσον αφορά τον θεμητό ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε το ότι οι ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές επενδύσεων να μπορούν να είναι σε ανταγωνισμό με φορεί που υπόκεινται σε κανόνε παρεμφέρεις παρομοίου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις απαιτήσει της θεμελιώδης που υπάρχουν και που προβλέπονται στο ΜΙΦΙΔ και ΜΙΦΙΡ. Το δεύτερο σημείο αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα Εν αυτή τη ενία οι τροποποίησεις ε, που έλαβαν χώρα από τον εισηγητή για καλύτερη πλαισίωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν επενδυτικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών ε, κατά την άποψή μου είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μπέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ συμπληρώνοντας αυτά που είπε και ο ιτρία κύριε Ντελφό, ε, με τα οποία συμφωνώ εν γέννη, θα ήθελα να αναφερθώ εκ νέου ε, στο θέμα του των τριών κατηγοριών των φορέων αυτών, των εταιριών και να αναφέρω μια μέρημνα που υπάρχει που προσπάθησε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ειδικό καθεστώς για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει σύγχυση με δραστηριότητα τύπου ιονή τραπεζική, θα πρέπει να βρούμε ε, να θεσπίσουμε παρόμοιες απαιτήσεις όπως αυτές που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες σεβόμενη την αρχή της ε, αναλογικότητας και να, αν έχουμε τρεις κατηγορίες τέτοιων φορέων και μπορεί να υπάρχει μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο βέβαια, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, να υπάρχει απέτηση κάθε φορέα που μοιάζει με τράπεζα ή που ασκεί δραστηριότητα ιονή τραπεζική, να μην μπορεί να ωφελείται από ένα καθεστώ πλέον ευνοϊκό που θα υπονόμευε και τη βάση του ανταγωνισμού και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις ε, διατάξεις, τις σχετικές με τις αμοιβέ Άκουσα αυτό που είπε ένα συνάδελφο, ο κ. Λούκα νομίζω που παρενέβη από αυτού. Θεωρώ ότι οι διατάξει για τι αμοιβέ και του μισθού είναι ένα στοιχείο ιονή ε, συστημικό, αν μπορώ να το πω αυτό, ε, του όλου διατακτικού, διότι γνωρίζουμε τι παρεκκλήσει που μπορεί να λάβουν χώρα στον τομέα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τι ε, αντιστοιχεί ισοδυναμίε, εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε δυσκολία. Βλέποντα κάποιε τροπολογίε του εισηγητή, βλέπω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Ποιος είναι αυτός. Μέσω της εκθέσεως να προδικάσουμε τη λύση που θα καθορίσουμε σαν Οικονομική Νοσηματική Επιτροπή για το καθεστώς των ισοδυναμιών στην έκθεση Hayes. Και ο κ. είπε ότι σε κάποιο στάδιο ίσως το καθεστώς ισοδυναμίας να χρειαζόταν πολιτική ε, διαμεσολάβηση και αναφερθήκατε στην ισοδυναμία με την Ελβετία στο τομέα Μιφίντ Μιφίρ. Όλη η συζήτηση που διεξήχθη, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταδεικνύει ότι αντιθέτως ένα στέρεο καθεστώς ισοδυναμίας εδράζεται επί τεχνικής αξιολόγησης. Αξιολόγησης των προτύπων που εφαρμόζεται από τις διάφορες πλευρές. Και αυτό σχετίζεται με μια μονομερή εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν πούμε ότι αν εξαρτάται από άμεση παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου και από συναπόφαση ισοδυναμία, προδικάζουμε απόλυτα το καθεστώς ισοδυναμίας που θα καθορίσουμε μετά την εξέταση της εκθέσεως Brian Hayes και νομίζω ότι υπάρχει ένα μεθοδολογικό πρόβλημα. Πώ αποφασίζουμε για τη συνοδυναμία που θα εφαρμόσουμε εδώ χωρί να έχουμε συμφωνήσει εν γέννη στα πλαίσια τη εκθέσεω του Brian Hayes και μετά επί τη ε, ουσία για το καθεστώ της ισοδυναμία πρέπει να είμαστε πολύ στεναροί όσον αφορά το καθεστώ. Δεν θέλουμε να καταστήσουμε έφταστη την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ούτε όπως είπε ο εισηγητής να δώσουμε στους απ' έξω ένα, μια προνομιούχα θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ένα καλό σύστημα ισοδυναμίας, καλά καθορισμένο, που θα, θα είναι αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε μετά τη σωστή συζήτηση της εκθέσεως του Brian Hayes. Για μας το θέμα της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών και εξετάσεως της εκθέσεως, ανεξάρτητα από το ρυθμό του Συμβουλίου, είναι σημαντικό. Καμιά φορά το Συμβούλιο πάει πιο γρήγορα από εμά, καμιά φορά πολύ πιο αργά, πολύ πιο συχνά πάει πιο σιγά από εμά. Αν κατ' εξαίρεση προχωρήσει πιο γρήγορα από εμά, επ' αυτού πιστεύω ότι η συνοχή και η λογική επιτάσσουν να διαθέσουμε, να δώσουμε σε αυτού μας περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε ένα το σημαντικό θέμα ε, και στο γενικότερο πλαίσιο του Brexit. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό τη επιτροπή μα, άλλωστε, να βρίσκουμε τη σωστή ισορροπία. την παρέμβασή σα. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας λάβει το λόγο, αν αυτό επιθυμεί βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σιγητά εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συζήτηση και για την υποστήριξη που παρατήρησα μέσω της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αποτελεί ενθάρρυνση για μας. Για μένα είναι ευκαιρία να επενθυμίσω ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέλαμε να επιδιώξουμε στο κείμενο. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η ποικιλομορφία των επενδυτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χρηματοδοτική αγορά τη Ευρώπη, να υπόκειται σε κανόνε προληπτικού που καλύπτουν πραγματικά του κινδύνου που δημιουργούν. Αυτό δεν νομίζουμε ότι ισχύει τώρα διότι το νομικό πλαίσιο που καλύπτει αυτές τις επιχειρήσεις πνίγεται στο νομικό πλαίσιο που αρχικά είχε δημιουργηθεί για τις τράπεζες. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε μέσω του κειμένου ήταν πραγματικά να εντοπίσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν αυτές οι εταιρείε και να τις θέσουμε στις απαιτήσει κεφαλουχικές που είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες και αφορούν τους συγκεκριμένους κινδύνους. Τι ο τρόπος θέλαμε να πετύχουμε έναν άλλο στόχο ένα στόχο απλούστευση και αναλογικότητα, διότι αναγνωρίζουμε επίση ότι αυτέ οι επιχειρήσει παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τι μεταπιστικές αγορέ τη Ευρώπη και χρηματοδότηση της οικονομίας και θεωρήσαμε χρήσιμο να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνε που θα του επιβάλλουμε θα του επιτρέψουν να συνεχίσουν να παίζουν αυτό το ρόλο, να κάνουν αυτή τη δουλειά, βέβαια όμω ταυτόχρονα να υπόκειται σε προληπτικέ προδιαγραφέ κατάλληλε. Ε, τρίτος ο οποίο συζητήθηκε επίση σήμερα και ήταν και δικό μα στόχο να εξασφαλίσουμε ότι το καθεστώ που θα εφερμόσουμε στις επιχειρήσεις των χωρών να είναι καθεστώς ενισχυμένο, λαμβάνοντα υπόψη ότι ιδιαίτερα οι κανόνες ισοδυναμίες που υπάρχουν σήμερα ε, συνελήφθησαν σε μια εποχή, σχεδιάστηκαν σε μια εποχή όπου οι προπτικές να έχουμε υπηρεσίες που παρέχονται από χώρες, από, από, από τρίτες χώρες ήταν λιγότερο σημαντικές από ότι αυτό που γινόταν στο εσωτερικό. Και γι' αυτό με αυτή την πρότασή μας Θέλαμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσει οδυναμίας για τις τρίτε χώρε. Αυτές που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς το κάναμε αυτό, Επεκτείνοντας τους κανόνες αναφοράς για να λαμβάνονται οι αποφάσει περί ισοδυναμία, ούτως ώστε να υπάρχουν οι κανόνε κοινοί στο βαθμό του δυνατού όσον αφορά τους κανόνε που εφαρμόζονται για τις τρίτε χώρε και τους κανόνε που εφαρμόζονται εντό Ευρώπη, αλλά θέλαμε να εξασφαλίσουμε και το ότι οι διαδικασίες και οι έλεγχοι, η εποπτεία εκ των υστέρων θα ενισχυθούν και θα εξασφαλίζουν ότι θα επιτυγχάνουν πραγματικά ισότιμους κανόνους παιχνιδιού μεταξύ των ευρωπαϊκών παρόχων και των παρόχων τρίτων χωρών. Σημειώσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις τροπολογίων που υπευλήθησαν από τον συγκητή. Πιστεύω ότι καλύπτουν ευρέω ε, τα σημεία που ανέφερα και βέβαια είμαστε στη διάθεση ε, του εισηγητού και της Επιτροπής σας, ούτως ώστε να σας βοηθήσουμε και να συμμετάσχουμε για την εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για αυτά τα ζητήματα. Κάτι τελευταίο, διότι ο κύριος Γκίγκολτ μας έθεσε μια ερώτηση, πιστεύω, όσον αφορά τους asset managers, πώς καλύπτονται οι asset managers στην πρόταση. Πράγματι, αληθεύει ότι η προσέγγιση που ακολουθήσαμε όσον αφορά την ταξινόμηση εν γέννη είναι ποσοτικής φύσεως. Θέλω να δούμε το μέγεθος των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται αυτοί οι φορείς και συναρτήσει του μεγέθους των δραστηριοτήτων να τους βάλουμε στην κατηγορία 2 ή 3. Αλλά δεν είναι μόνο ποσοτική προσέγγιση, αλλά και ποιοτική. Διότι θέλαμε μέσω της πρότασης, όπως κάνουμε για τον ορισμό των επιχειρήσεων που είναι συστημικές ουσιαστικά θέλαμε να δούμε να εντοπίσουμε κάποια είδη υπηρεσιών που θεωρήσαμε που δικαιολογούν να αντιμετωπιστούν με τρόπο πιο προληπτικό, πιο προσεκτικό από ό,τι άλλες δραστηριότητε όπως είναι το trading. Στο πλαίσιο αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι το τρόπος ότι αυτές οι δραστηριότητε του trading να ασκούνται σε επίπεδα υψηλά και σε επίπεδο συστημικό. Και εδώ απαντώ και σε αυτά που μας ε, είπε η κυρία Μπέρες στην παρέμβασή σας. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τράπεζες. Να υπάρχει ένα επίπεδο σύγκλησης των κανόνων και να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός στο βαθμό του δυνατού σε αυτούς τους τομείς. Αυτά ήθελα να πω. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ για τις θετικές αντιδράσεις της Επιτροπής σας όσον αφορά την πρότασή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας κύριε Σιγητά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις. Και τώρα να στραφούμε στον κύριο Φέρμπερ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές παρατηρήσεις. Αποδεικνύουν ότι σε ορισμένα σημεία θα συμφωνήσουμε σύντομα, ενώ σε άλλα σημεία χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό για τέτοια θέματα. Τονίζω ότι εκπλήσωμαι για ορισμένα από αυτά που άκουσα. Πρώτα απ' όλα από την αρχή είχα στείλει το χρονοδιάγραμμα συναντήσεων στους σκιώδες αλλά εγώ επιπλέον τήρησα αυτό το χρονοδιάγραμμα με βάση τις προθεσμίες που είχα ο ίδιος θέσει έστειλα την έκθεσή μου για μετάφραση αυτό ίσως να εξέπληξε ορισμένου. Κανείς δεν υπέβαλε αντιρρήσεις για αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ε, ε, τώρα επίσης με εκπλήσει το ότι άκουσα ότι θα πρέπει να υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας για να καθορίσουμε ορισμένα θέματα και συγκεκριμένα το θέμα των ε, ισοδυναμιών. Τότε δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση Χιούμπνερ που έχει συγκεκριμένη σημασία. Θα πρέπει να την περιμένουμε. Ή θα ψηφίσουμε για όλες τις εκθέσεις είτε για καμία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να γίνει για το ίδιο θέμα σε μία έκθεση και κάτι δεν μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και κατόπιν θα αξιοποιήσουμε και αυτά που θα προκύψουν από την έκθεση Χάις. Στην έκθεση Χιούμπνερ δεν ξέρουμε ακόμη τι θα περιληφθεί για την ισοδυναμία. Ανέφερα το παράδειγμα την Ελβετία, αλλά αγαπητοί υπερβάνους θα μπορούσα να αναφέρω και τη ΣΥΠΑ. Εδώ συμφωνήσαμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που προτείνει η Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και χωρίς να έχουμε δικαίωμα στην απόφαση, επιτύχαμε η ισοδυναμία αυτή να περιοριστεί σημαντικά για να μην δημιουργηθούν κενά μέσω των οποίων μικρέ μικρές ε, αγορές αξιογράφων των Ηνωμένων να επηρεάσουν τις δικές μας ε, αγορές χειρογράφων. Και από ό,τι θυμάμαι, συμφωνούσαν οι σοσιαλιστές με αυτό. Ανέφερα άλλο παράδειγμα, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω και αυτό που μόλις ανέφερα. Τρίτον, οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες θα παραμείνουν στο καθεστώς CRD. Δεν το αλλάζει αυτό η έκθεσή μου. Δηλαδή, Γι' αυτό που λέμε για τις δημόσιες αναχώρα εκθέσεις, η υποχρέωση γνωστοποίησης των δεδομένων τους για τις αμοιβέ των στελεχών τους. Όλα αυτά θα παραμείνουν. Το θέμα όμως είναι αναλογικότητα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια επενδυτική εταιρεία ε, δισεκατομμυρίων με τον ίδιο τρόπο με μια επενδυτική εταιρεία λίγων εκατομμυρίων. Και ανέφερα περισσότερο και το θέμα της συστημικής σημασίας. Πού μπορούμε να ελαφρώσουμε με βάση, να ελαφρύνουμε με βάση την ε, αναλογικότητα και χωρίς να υπάρχει αύξηση των κινδύνων την κατάσταση. Αυτός είναι ο προσανατολισμός μου και θα ήθελα να συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε. Για την τροπολογία 28 έχω αναφέρει πολλά στο σχέδιο έκθεσης ε, που την αιτιολογούν. Δεν θέλω οι επενδυτικές εταιρείε τρίτων χωρών να αντιμετωπίζονται καλύτερα από τις δικές μας. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν πράγματα που απαγορεύονται στι δικέ μα εταιρείε. Πρέπει να το συζητήσουμε. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, τότε στην περαιτέρω συζήτηση να το δούμε. Όμω, εγώ δεν συμφωνώ. Κάτι τέτοιο θα πήγαινε εντελώ προ την αντίθετη κατεύθυνση. Όσα δεν επιτρέπονται σε εμά, δεν μπορούν να επιτρέπονται σε τρίτου. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Γιατί αλλιώ θα φύγουν όλε οι εταιρείε αυτέ από την Ένωση. Και οι δυνατότητε ε, προληπτικής ε, αντιμετώπιση και ελέγχου των εταιριών τρίτων χωρών θα είναι <clears throat> ελάχιστες. Είμαι ανοιχτό προ συζήτηση, εγώ είμαι αντίθετος, αλλά αν η πλειοψηφία θέλει κάτι άλλο, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται ανάγκη διευκρίνηση. Πρέπει να κάνουμε μια σειρά συναντήσεις των σκιωδών για να διευκρινίσουμε την κατάσταση ανεξάρτητα από τι προθεσμίε για τι τροπολογίε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Διότι εάν δεν καθορίσουμε την προθεσμία για τι τροπολογίε, δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιώδη συζητήσει. Πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση με ένα λογικό ρυθμό. Να μην τα αναβάλουμε όλα για μήνε. Εντάξει, θα μπορούσα να συμφωνήσω για να ε, επιμηκυνθεί η προθεσμία μια-δύο εβδομάδες, αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να συζητήσουμε με να επιτύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συμβαστικές λύσεις, γιατί κατόπιν ε, θα έρθουν οι διακοπές. Αν αρχίσουμε τους τριμερείς διαλόγους μόνο τέλη του χρόνου, δεν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος της θητείας. Γιατί θεωρώ και γι' αυτό έκανα τόσο γρήγορα την έκθεσή μου, θεωρώ ότι έχουμε μια ρεαλιστική, ρεαλιστική πιθανότητα να προλάβουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό πριν τη λήξη της θητείας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παρά όλες τις διαφορετικές απόψεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε να περάσει το θέμα αυτό στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάρκους. Συνοψίζω. Α, παρακαλώ. Συγγνώμη που παρεμβαίνω εκ νέου, κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα της προθεσμίας για τις τροπολογίες, καταλαβαίνω, αλλά υπενθυμίζω, ότι ο πρόεδρος καθορίζει τις ε, προθεσμίες και όχι ο εισηγητής. Ο πρόεδρος καθορίζει με βάση τις προτάσεις του εισηγητή. Δηλαδή, μουτάτης μουτάντης, αυτά που γίνονται στην Ολομέλεια, γίνονται και εδώ στις Επιτροπές. Σημειώνω ότι τα επιχειρήματα για την ταχύτητα των συζητήσεων και για το πότε θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό είναι απόλυτα σωστά. Θέλω να ολοκληρωθεί η συζήτηση πριν τη λήξη της θητείας. Αλλά Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δεν θα τα αναφέρω. Θα θυμάστε σε τι ε, αναφέρομαι. Όπου θέλουμε να ολοκληρώσουμε και αυτά τα θέματα εντός της ζητίας αλλά είναι πολύ πιο γενναιόδωρο το χρονοδιάγραμμα. Οπότε θα πρότεινα να αναφερθείτε στον πρόεδρό μας, στον πρόεδρο της Επιτροπής, για να υπάρξει δυνατότητα να αναβληθεί για ένα μήνα να παραταθεί για ένα μήνα η προθεσμία της τροπολογίας. Για τα, όπου συμφων... για τα σημεία όπου συμφωνούμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για να εξετάσουμε τις διάφορες ισοδυναμίες που είναι θεμελιώδες θέμα δεν είναι δυνατόν ότι μπορούμε να αποφασίσουμε εάν δεν κάνουμε μια πρώτη συζήτηση ως Επιτροπή για την έκθεση Hayes. Κύριε Σιγητά, λοιπόν, Και ε, τελικά απευθύνομαι σε εσά κύριε Πρόεδρε να μην ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό σήμερα, να λάβετε υπόψη το αίτημα, το ιδιαίτερα έντονο αίτημα των σοσιαλιστών της ομάδας μου να παραταθεί για να μην είναι προθεσμή για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να... Κάνουμε μια σύνοψη λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα τροπολογίες 24 Μαΐου μεσημέρι συζήτηση 18 Ιουνίου, 24 ψηφοφορία Σεπτεμβρίου και το η Ολομέλεια θα ψηφιστεί εκεί. Να πω ότι δεδομένων των συνθήκων ζητώ από τον κύριο Γκουαλτιέρη που είναι πρόεδρος να μπει σε μια συζήτηση με τον εισηγητή και τους εκπροσώπους αυτής της πρότασης και να εξετάσει όλα τα εναλλακτικά σενάρια έτσι ώστε να διευκρινιστεί και το θέμα του χρονοδιαγράμματος της Προεδρίας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως έχουμε ε, τη δυνατότητα το φάκελο αυτό να τον οδηγήσουμε σε επιτυχημένη λύση το συντομότερο δυνατόν. Κύριε Φάρμπερ, κύριε Γκολτιέρη και εσείς ε, δείτε το θέμα αυτό για να βρείτε ποια είναι η καλύτερη λύση. Πάντως ε, προς το παρόν θα ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα όσο έχει. Σίγουρα ο κύριος Γκουαλτιέρη θα μας ενημερώσει το συντομότερο. Σας ευχαριστώ.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 Υπότιτλοι it Καλώ ήρθατε συνάδελφοι, πολύ σημαντική ψηφοφορία, όπως ξέρετε θα ψηφίσουμε δύο σημαντικές εκθέσεις για δύο κανονισμούς στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου για την Ένωση των Κεφαλαγορών, η αγορά και τον αντίκτυπο που θα έχουν κάποια γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Παρακαλώ λοιπόν να κάνουμε μια δοκιμή καταρχήν των μηχανημάτων. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας να ψηφίσετε. μπορούμε να ξεκινήσουμε με την έκθεση Langen για το Refit τροπολογία 77-79 υπέρ κατά εγκρίνεται ας γίνει έλεγχος ξεκινάει ο ηλεκτρονικός έλεγχος Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 καταπίπτει. Συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε ξεχωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 80 για τη μερική ε, έγκριση κάποιων λέξεων στον κατάλογο ψηφοφοριών. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το τροπολογία 121 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρας απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123, 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 125 υπέρ κατά έλεγχος όλοι οι φιλεύθεροι είναι υπέρ γίνει έλεγχος άρχεται πέρας Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τοπολογία 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μια ψήφος 176 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά ψηφ... ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 5, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5α. Καταπίπτει. Πάμε στην 188 λοιπόν. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Θα ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν μπορούσα να δω όλα τα χέρια. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Πέρας. Ναι, πραγματικά απορρίπτεται. 190, 190 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με την ίδια διαφορά ψήφων 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203-204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 218-219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 11 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 254. Χορήγεται μόνιμη εξαίρεση από τα ΙΕΝΣΕΙΣ υπέρ. Αυτό το τμήμα. Υπέρ. Είσαστε κατά νομίζω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.75 και 2.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ετελογική σκέψη 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά απο... έλεγχος για την 34 άρχεται Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. «41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο που τροποποίησαμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας 46 ψήφοι υπέρ 4 ψήφοι εναντίον 5 εναντίον μάλλον και 4 αποχές οπότε το κείμενο του ψηφίσματος εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η πρόθεσή σας για το επόμενο στάδιο. το ΕΛΚ προτείνει να συντηρηθεί στην Ολομέλεια. Ο συζητητής στηρίζω το αίτημα αυτό και να μην ψηφίσουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων, να απορρίψουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Μα... Δεν υπάρχει αίτημα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.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 αποχές εγκρίνεται. 467 και 473 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 468 και 472 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 469 και 471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 474 474 4,74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 501 γιατί νομίζω εδώ έχουμε κάποιο λάθος στον κατάλογο Α, έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 504 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 505 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 554 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 555 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 569 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 570 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 576 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 577 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 578 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 37 υπέρ κατά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 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικά την 114 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 140 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 140 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική 43 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 170, 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 45 υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα λοιπόν, ονομαστικά, έχουμε τελειώσει πρόεδρε. Όχι, τώρα ονομαστικά θα γίνει η ψηφοφορία ονομαστική για την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων επί τη βάση της έκθεσης που μόλις εγκρίθηκε, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. 47 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές, οπότε και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μια υπαρκέστατη ε, πλειοψηφία. Κύριε Λάμπερτς, κύριε Πρόεδρε, Τώρα που σας άκουγα και επειδή δεν θα ήσασταν ο πρόεδρος της ΕΚΟΝ ε, την επόμενη θητεία να γίνεται πρόεδρος της, ε, του Κοινοβουλίου γιατί τόσο καλά που τα πήγατε θα ήταν υπέροχα και αν κάνατε και ένα διαγωνισμό με τον κύριο Βίλαντ να έχετε τον ίδιο κατάλογο ψηφοφοριών και να κάνουμε ένα διαγωνισμό ποιος θα τα πει πιο γρήγορα γιατί νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα τεράστιο αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος, θα το σκεφτώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Αύριο θα ξεκινήσουμε και πριν το πω αυτό θα ήθελα καταρχήν να σας πω πως είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τόσο μεγάλη πλειοψηφία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ε, γκρίναμε τόσο δύο τόσο σημαντικές εκθέσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητέ για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που κάναμε. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα πολύ δυνατό ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δείξει το δρόμο στο Συμβούλιο και να προχωρήσει ε, με φακέλου σημαντικούς πολύ γρήγορα για την χρηματοσπιτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στους εισηγητέ και σε όσους είχαν αναλάβει ε, κομμάτι αυτού του φακέλου. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9